Goedemorgen Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα να προεδρεύσω σήμερα το πρωί τη συνεδρίασή μας. Έχετε μπροστά την ημερήσια διάταξη όπως ανακοινώσαμε ήδη την Τρίτη, πρέπει να προσθέσουμε ένα σημείο εδώ. Έτσι αποφασίσανε οι συντονιστές στη συνεδρίασή τους. Μετά τη συζήτηση που κάναμε για την απαλλαγή και την ε, συνέχεια που θα δώσουμε στην υπόθεση ΣΕΠΟΛ, αποφασίσαμε να προσθεθεί και αυτό το σημείο. Προτείνω λοιπόν να το βάλουμε σημείο 2β, δηλαδή ανάμεσα στις ανακοινώσεις του Προέδρου και την συζήτηση της ε, έκθεσης Καταλήν Τσόριν Ιβάνου. Συμφωνείτε? Γιατί πρέπει μετά να ψηφιστεί στην ε, Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, την πρώτη, τη δεύτερη, θα δούμε. Συμφωνείτε λοιπόν με την τροποποίηση αυτή στην ημερήσια διάταξη. Καλώς. Έχω δύο ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτον, χθε το απόγευμα, το βράδυ, πήραμε μια επιστολή από τον επικεφαλής της μονάδας που είναι υπεύθυνο ε, για την τηλεόραση Europarla. Το ξέρετε ότι είχαμε ρωτήσει τον Κλάους Βέλε και μετά από συζήτηση με την Αντιπρόεδρο Κράτσα, η Europarl TV ζητάει στα πλαίσια της απαλλαγής επίσης σε σχέση με τον προπολογισμό, έκθεση Ιτάλα, θα ήθελε να συναντηθούμε με τους εκπροσώπους και η Αντιπρόεδρος Κράτσα λέει στο Στρασβούργο να γίνει αυτό στις 16 Φεβρουαρίου. Τετάρτη στο Στρασβούργο. Κάποια συγκεκριμένη στιγμή που θα δούμε ποια θα είναι αυτή. Μια συνάντηση, θα προσκληθείτε κι εσείς. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει διερμηνία, θα είναι στα αγγλικά αυτή η συνάντηση μαζί τους. Θα σα σταλούν οι προσκλήσει πάντως για την τη συνάντηση αυτή με τους ανθρώπους της Europarla για να ενημερωθούμε εν ώψη της ε, απαλλαγής που μελετάμε. Δεύτερον, συνάντηση συντονιστών που έγινε την Τρίτη το βράδυ. 5.30 με 6.30. Πήραμε πολλές αποφάσεις. Η σε διάταξη ήταν πυκνή. Υπάρχουν πάντω τα πρακτικά με την απόφαση των συντονιστών. Σήμερα το απόγευμα μάλλον θα είναι έτοιμο και θα σας ταλούν. Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένες οι αποφάσεις των συντονιστών. Εφόσον δεν θα μας πείτε τίποτα για αυτές. Σέπολ τώρα, κλείσιμο λογαριασμών. Το σημείο που προσθέσαμε. Εδώ έχουμε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει έρθει που μιλάει για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κλείσιμο των λογαριασμών για το 2008. Η Βερονίκ Ματιέ είναι η συγκήτρια. Κύριε Ματιέ, έχετε κάτι να πείτε Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση του κυρίου Ντί. Αν συμφωνείτε κι εσείς θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ντί για να μας εξηγήσει γιατί προτείνει αυτή την προφορική τροποποίηση. Μετά θα δώσω σε εσά το λόγο για να μας πείτε τη δικιά σας άποψη και μετά πρέπει να ζητήσω ε, από τους αδέρφους να μου πούνε κατά πόσο συμφωνούν να θέσουμε σε ψηφοφορία την προφορική τροποποίηση. Αν όλοι συμφωνείτε, εντάξει, αν δεν συμφωνείτε, δεν γίνεται. Αν συμφωνείτε θα την ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε δηλαδή την τροπολογία με την προφορική τροποποίηση. Ο κύριος Σοντή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι μεταξύ εκείνων των βουλευτών που θεωρούν ότι θα πρέπει να κλείσουν το ταχύτερο δυνατό οι λογαριασμοί. Θα ήθελα να προτείνω ε, η λέξη approve, εγκρίνει, που δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να εννοούμε ότι εγκρίνουμε λογαριασμούς, γιατί εδώ ξέρουμε ότι είναι εσφαλμένα τα στοιχεία του 2008, οι λογαριασμοί δηλαδή, και ότι η διόρθωση δεν έχει γίνει με βάση διορθωμένους λογαριασμούς 2008, αλλά με βάση διορθωμένους λογαριασμούς 2009 με 1,2 και 1,4 εκατομμύρια ευρώ διόρθωση. Ως εκ τούτου λοιπόν η πρότασή μου, η οποία εντάσσεται στο άρθρο 5 της παραγράφου 6 του ιστορικού μας κανονισμού, γιατί όταν υπάρχει αναβολή για λόγους ε, άρνησης, κατά τη διαδικασία της απαλλαγής, μπορούμε να ζητήσουμε από το Κοινοβούλιο την τυπική, ε, το τυπικό κλείσιμο της υπόθεσης. Αν λέγαμε λοιπόν το approve θα μπορούσε να παρερμηνευτεί αυτό ως ε, ότι εγκρίνουμε τους λογαριασμού, πράγμα το οποίο βέβαια δεν εννοούμε. Και γι' αυτό ε, θα έλεγα η λέξη approve να αντικατασταθεί με το decide. Αποφασίζει το κλείσιμο των λογαριασμών. Ευχαριστώ η κυρία Ματσιό, η Για να αντικαταστήσουμε στην παράγραφο 1, αυτή είναι η πρόταση δηλαδή, το approves με το decides. Αντί για εγκρίνει, αποφασίζει δηλαδή. Κυρία Ματιέ, τι λέτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά το δέχομαι. Δεδομένου ότι το σημαντικό εδώ είναι να κλείσουμε τους λογαριασμούς. Είμαι υπέρ λοιπόν της ε, τροπολογίας. Θα ήθελα ωστόσο να διευκρινίσω πως ε, καθυστέρησα προ το κλείσιμο των λογαριασμών και με πολύ μεγάλη χαρά τους κλείνω σήμερα. Αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα για τα οποία δεν θα είχαμε λάβει γνώση εάν είχαμε κλείσει νωρίτερα τους λογαριασμούς και ιδιαίτερα στα διορθωτικά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Οντί νωρίτερα, καθώς και το γεγονός ότι ο νέος ε, διευθυντής, ο κύριος Μπόμφη, μάλλον τα όσα μας είπε ο κύριος Μπόμφη, ο νέος διευθυντής δηλαδή. Και θα ήθελα να επαναλάβω ότι δέχομαι την πρόταση του κύριου Όντι. Ε, Σας ευχαριστώ. Ωραία. Τότε ρωτάω, έχει κανείς αντίρρηση να ψηφίσουμε αυτήν την προφορική τροποποίηση. Γιάννης. Ως προς το περιεχόμενο δεν έχω αντίρρηση. Συμφωνώ με τον κύριο Οντζή. Θα έλεγα όμως για το αγγλικό κείμενο μήπως το to agree, συμφωνεί, αντί για το decide, είναι καλύτερο. Συντακτικά μόνο η διόρθωση. Ότι τι λέτε. Ναι, θα ήθελα να πω ότι το γεγονός... Να επαναλάβω την ε, ε, συλλογιστική μου. Εάν πούμε τη λέξη agrees, συμφωνεί, θα δοθεί εντύπωση ότι συμφωνούμε με τους λογαριασμούς. Το πρόβλημα είναι ότι οι λογαριασμοί 2008 είναι σφαλμένοι. Αν δεν σας κάνει το αποφασίζει, decide, decides, να πούμε κλείνει τους λογαριασμούς. Το κοινοβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς. Αντί αποφασίζει να κλείσει, Κλείνει του λογαριασμού, να μην βάλουμε δηλαδή ε, κύριο ρήμα. Κλείνει του λογαριασμού. Ε, με, αυτή την τελευταία παρατήρηση του κύριου Ντί συμφωνείτε. Μπορείτε δηλαδή να συμφωνήσετε να ψηφίσουμε. Κλείνει τους λογαριασμούς. Απλά και μόνο. Και τίποτα άλλο. Η συγκίτρια συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερη διατύπωση αυτή. Πρόεδρος, καλώς. Τότε θα ψηφίσουμε με τις κάρτες σας παρακαλώ. Ε. Έχετε τις κάρτες σας μαζί. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Ξεκινάει, αρχίζει μάλλον η ψηφοφορία. Με μετρήσουμε έτσι νομίζω ότι θα φανεί. Καθένας είναι υπεύθυνο. Ψηφίστε. Μην καθυστερείτε. Η συγκίτρια, εντάξει, είναι έτοιμη. Ωραία. Ωραία. Ψηφίζουμε και το αποτέλεσμα είναι 18. Ψήφισαν 18 υπέρ, κανείς κατά, κανείς αποχή. Ομόφωνα λοιπόν. Οπότε συγχαρητήρια και συγχαρητήρια κύριε Οντή και την κυρία Ματιέ βέβαια για τη δουλειά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, τα καταφέραμε. Ξέρω ότι η εμπειρία ήταν δύσκολη, τώρα και ο κύριος Σταυρακάκης βέβαια αναλαμβάνει. Ελπίζω να μην επαναληφθούν τα δυσάρεστα. Φτάνουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Είναι η ετήσια έκθεση 2009. Η συγκέντρια είναι η Καταλήνη Σόριν Ήβαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Ιβαν, ο κύριος Καταλήν Σόριν Ιβαν. Κύριε Πρόεδρε, είχα ετοιμάσει την παρουσίασή μου στα ρουμανικά για σήμερα, αλλά για σήμερα δεν είναι επίσημη γλώσσα. Δεν περιλαμβάνεται στο γλωσσικό καθεστώ στα ρουμάνικα. Θα μιλήσω λοιπόν αγγλικά. Θα κάνω μια πιο σύντομη παρουσίαση και δεν θα περιλαμβάνει και τόσες λεπτομέρειες ε, θα σας έδινα πολύ περισσότερη στη μητρική μου γλώσσα, στα ρουμανικά. Ακούω ότι προσπαθούν να βρουν μια λύση ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε ρουμανικά και να μεταφραστούν τα ρουμανικά. Οπότε από τη στιγμή που θα έχει λυθεί το πρόβλημα, γιατί αυτό μου λένε τώρα από την Ολλανδική καμπίνα, μόλις έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα θα ενημερωθείτε και θα μπορέσετε να μιλήσετε ρουμανικά τότε από εκείνη τη στιγμή, εντάξει. Εντάξει, γιατί στις 10 πρέπει να μεταβώ σε μια άλλη συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μεγάλες πιέσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όχι μόνο γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τη χρηματοοικονομική κρίση, αλλά και γιατί οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είναι διατεθειμένες να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παρά το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν περισσότερες προτεραιότητες ε, στο πρόγραμμά μας μετά από την ε, θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Να πω εν συντομία ότι θα ήθελα να συγχαρώ την Όλαφ ε, για τις δραστηριότητές της. Πρέπει να πω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από πλευράς τους είναι ο πιο σημαντικός οργανισμός στην καταπολέμηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια θα πρέπει να πω ότι αυτό δεν αρκεί. Μεγάλο μέρος της ευθύνης βαραίνει τα κράτη-μέλη και δεν γίνεται εξίσου καλή δουλειά με την Όλαφ. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες σε εθνικό επίπεδο Και θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πιέσει περισσότερο τις ε, εθνικές κυβερνήσεις Για τους ίδιους πόρους υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, όπως ε, αποδεικνύεται από το ελεγκτικό συνέδριο για τις ε, διατάξεις των εθνικών τελωνιακών κυρίως για τις επιλογές των εμπεριβομένων και τις εισαγωγές και το ποιοι θα ελέγχονται στα τελωνία. Πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την εποπτεία τους στα τελωνία και να ενισχύσουν και τα συστήματα τελωνία ώστε να υπάρχει και κατάλληλη υποστήριξη. Είναι ζωτική σημασία να υπάρχει μια σαφής και συγκεκριμένη εικόνα προτού αρχίσουμε να εξερευνούμε πιθανέ λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν σαφέστερα, πιο αξιόπιστα και πιο συγκρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εξακολουθούν να διαπιστώνονται προβλήματα Κάποια κράτη-μέλη δεν παρέχουν όλες τις πληροφορίες ε, ή δεν παρέχουν έγκαιρα τις πληροφορίες και σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές ε, δεν είναι εύκολα συγκρίσιμες. Για τις δαπάνες στο γεωργικό τομέα, Τα ευχάριστα νέα είναι ότι βελτιώθηκε το σύστημα αναφορών στον τομέα και πλέον έχουμε ε, σχεδόν 95% ε, στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν δίνουν τις εκθέσεις τους εγκαίρως, όπως για παράδειγμα η Αυστρία, η Φιλανδία, οι κάτω χώρες, η Σλοβακία και άλλες χώρες. Επιπλέον, διαπιστώνονται και προβλήματα κατά την εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ακούσαμε και τον Επίτροπο Τσόλος, ο οποίος ε, μίλησε για τη στρατηγική του προκειμένου να ενθαρρύνει τις χώρες αυτές να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή του συστήματος. Επιπλέον υπάρχει μια καταστροφική κατάσταση για το συνολικό ποσοστό ανάπτυξης σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Το 2009 είχαμε μόνο 42% από 1 δις 266 εκατομμύρια ευρώ είναι ελάχιστο το ποσό. Για την πολιτική συνοχής ε, υπάρχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα, αν όχι το σοβαρότερο πρόβλημα. Ε, το βασικό θέμα εδώ είναι η νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες. Ε, σε αυτό το τομέα θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η πρόοδος ταχύτερα για την ε, νομοθεσία, ε, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση. Είναι τελείως διαφορετικά τα συστήματα στα κράτη-μέλη, δεν είναι πάντα διάφανο το σύστημα και πολλοί οικονομικοί φορείς δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιους μειοδυτικούς διαγωνισμούς. υπάρχει και ειδικό πρόβλημα στο προς την πρόσβαση για τα γεωργικά θέματα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτή τη στιγμή βέβαια τα στοιχεία είναι αμφισβητούμενα, δεν ε, είναι σαφή. Έχω γράψει στην εκθεσή μου ότι οι βουλγαρικές αρχές δεν έχουν αναλάβει ε, επαρκή δράση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ποσοστό του 2% που αναφέρεται είναι αμφισβητούμενο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν. Έχουμε για άλλη μια φορά το ίδιο πρόβλημα που έχουμε με τις εκθέσεις από τα κράτη-μέλη και τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει ίσως να έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα εκθέσεων το οποίο να είναι πιο σαφές, πιο αξιόπιστο και να έχει και τη δυνατότητα σύγκρισης. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Ένα συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο, ο κύριος Βασίτης. Υπάρχει κανένα άλλο που θέλει το λόγο, θέλει κάτι να ρωτήσει. Ωραία. Μια στιγμή. Πρώτα, ίσω, καλύτερα θα ήταν να ακούσουμε τον κύριο Ήλιτς από την Όλαφ που έχει ζητήσει το λόγο για να μα ενημερώσει. Οπότε καλύτερα να μα μιλήσει πρώτα ο κύριο Ήλιτ και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέρφους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως ήταν σκόπιμο να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν μου ξαναδώσετε το λόγο στερα από αυτά που σκοπεύω να πω Πρόεδρε δεν θα εκπροσωπώ την όλα, αλλά ολόκληρη την Επιτροπή. Γιατί χρειάζεται να καλύψω κάποια θέματα που υπαγόνται σε αρμοδιότητες και άλλων υπηρεσιών τη επιτροπή. Μπορώ να συνεχίσω λοιπόν. Ευχαριστώ. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε για την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις ε, για το σχέδιο έκθεσης που είναι πολύ ενδιαφέρον και πιστεύουμε θα μας ε, βοηθήσει στο εγχείρημα στο οποίο έχουμε αποδειχθεί με τη βοήθεια βέβαια της Επιτροπής σας. Μια πρώτη και γενική παρατήρηση, ίσως σχετική και με προηγούμενες σχετικές ή συναφείς εκθέσεις της Επιτροπής σας. Ο εισηγητής έχει προφανώς σαφέστατη αντίληψη των ρόλων που διαδραματίζουν διάφοροι θεσμικοί παράγοντες αυτό που κάνει το ελεκτικό συνέδριο Φερρυπίν και ω εκ τούτου και οι εκθέσει που παράγει το ελεκτικό συνέδριο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνει η Όλαφ και ω εκ τούτου και από το περιεχόμενο των εκθέσεων τη Όλαφ. Εμεί προσπαθούμε εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό τη να ε, επιδοθούμε σε συλλογή και ανάλυση στοιχείων, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε πάρα πολύ αυστηρούς ε, κανόνες ε, διαδικαστικούς και ορισμούς, Φερρυπίν, για το τι σημαίνει παρατυπία. Ενώ το ελεγκτικό συνέδριο δεν περιορίζεται κατά αυτόν τον τρόπο και πολύ καλά κάνει, διότι έχει ε, ως μέθοδο αξιολόγησης κατάστασης μια επιστημονική, ε, βασισμένη δηλαδή σε επιστημονικά στοιχεία και αντικειμενική αξιολόγηση της ε, κατάστασης, της οικονομικής κατάστασης. Ασχολούμαστε και οι δύο με την οικονομική διάσταση των στρατιωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν ε, αλλά από διαφορετική σκοπιά και έτσι η διαφοροποίηση μπορεί να εμφανιστεί κατά καθοριστικό τρόπο, όπως φαίνεται και στην έκθεση που συζητάτε πολύ τώρα πιο συγκεκριμένα ο προσδιορισμός υποχρέωσης νομικού χαρακτήρα, δεσμευτικής δηλαδή υποχρέωσης για την ε, κοινοποίηση παρατυπιών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει, έχει προχωρήσει σε συνεργασία και με πολύ διάλογο με τα κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει αυτά τα συστήματα που λειτουργούν και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια τα σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης παρατυπιών, τα οποία έχουν φέρει ρηξικέλευτες αλλαγές, όχι μόνο ε, στον Ε, τρόπο με τον οποίο καταγράφονται παρατηρήσει, αλλά και στι δυνατότητε να περιοριστεί το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με αυτά. Και επίση έχουμε ε, ορίσει τη δυνατότητα μέσα από το παράρτημα στο, στην έκθεση του άρθρου 325 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της σχετικής ε, αναφοράς παρατυπιών και απατών στους διαφορούς τομείς που έχουμε μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να χαρτογραφήσουμε και πιστεύω ότι αυτές οι πληροφορίες και τα στοιχεία παρέχουμε είναι στατιστικά αποδεκτά και πιστεύω θα σας είναι χρήσιμο και στις συζητήσεις σας με τον εισηγητή. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε ε, δημοσία τουλάχιστον ε, ακριβής ή έστω κατά προσέγγιση πληροφορίες για το επίπεδο της απάτης. Είναι κάτι το οποίο εγώ αρνούμαι πάντοτε να πράξω δημόσια γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με, με εκτιμήσεις ως προς, την, ως μια εγκληματική δραστηριότητα πρέπει να είναι σαφές ότι μιλάμε για εκτιμήσεις μόνο και όχι για βεβαιότητες και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να αποφεύγουμε τη διάδοση πληροφοριών στο δημόσιο χώρο για ζητήματα τα οποία μπορεί να κρυθούν κατά διαφορετικό τρόπο ε, από άλλες αρχές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με υποχρεώνει να απέχω από την συζήτηση και τώρα και στο μέλλον. Για δε τα σχόλια ε, τα σχετικά με τα έσοδα της πράξης. που αν θέλετε, ε, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν βλάπτει τόσο το κύρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αλλά ταυτόχρονα είπε και ο εισηγητής ήδη είναι πολύ σημαντικό. Δεδομένων και των οικονομικών δυσχεριών που αντιμετωπίζει ένα του συνολότη αλλά και τα κράτη-μέλη επιμέρους. Για τους κανόνες σχετικούς με τις δημόσιες προμήθειες, είναι πιθανόν, για να το πω κομψά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πολύ πιθανόν μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει πράσινη βίβλο για το θέμα αυτό μέσα σε, στην προσεχή μια μισή ώρα. Αν είχα το λόγο λίγο αργότερα, ίσως θα μπορούσα να σας δώσω πιο πολλές πληροφορίες. Πάντως, θα δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, του πρωινού ακόμη, πρόοδο ως προς την υπόθεση αυτή. Αναμένεται βέβαια να αναπτυχθεί και βάση συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο πάντα την απλούστευση των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες και όταν έρθει η στιγμή και πάλι, δεν παραλαμβάνω, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια διατύπωση κατάλληλη, μια διατύπωση όπου και το γράμμα θα είναι ορθό αλλά και οι αρχές που ακολουθεί με βάση δηλαδή τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες σκοπεύουμε να ε, αποτρέψουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν και πάνω απ' όλα να διακρίνουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα τεχνικό σφάλμα από μια εγκληματική ή σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα σημαντικό αλλά και ευαίσθητο είναι οι κανόνε περί που στηρίζονται στην αρχή της συνένεση είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανεί την ανάκτηση σε ορίζοντα χρονικό σχετικά ευρύ διότι υπάρχουν βραδιπορίες ως προς τα προγράμματα. Τα προγράμματα έχουν κύκλους διαφορετικούς από, ε, από τον κύκλο του προϋπολογισμού και άρα η ανάκτηση έρχεται σε στιγμή πολλές φορές χρόνια μεταγενέστερη της πραγματικής δαπάνης. Και άρα είναι δύσκολο μερικές φορές ε, να έχουμε την συνολική θεώρηση και βέβαια και να ε, συναγάγουμε τα συμπεράσματα που θα έπρεπε και τα διδάγματα που θα έπρεπε από αυτή τη διαδικασία της ανάκτησης. Και εν τέλει, Πρόεδρε, ίσως στο θέμα του ποιες χώρες θα πρέπει να κατονομαστούν. Ε, δεν μπορώ βέβαια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προσωπώ εδώ να κάνω σχόλια σε λεπτομέρειες στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως αν μου επιτρέπετε να επισημάνω ότι θα ήταν ασφαλμένο να κατονομαστεί μόνο μία χώρα. Εάν με υποχρέωνε κανείς να δώσω κατάλογο των χωρών που θα πρέπει να κατονομαστούν, ασφαλώς δεν θα περιοριζόμουν μόνο σε μία. Θα, ήταν, θα επρόκειτο για πολλές χώρες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νέτ για τις πληροφορίες σας. Τώρα αν αργότερα θέλετε να πάρετε και πάλι το λόγο δεν έχετε παρά να μας το πείτε. Πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Βασίτης, ο κύριος Ντόιτς, ο κύριος Σάντεργκαρτς, ο ε, κύριος Γκάιερ, την κυρία Μακοβέη και εσείς επίσης, συνάδελφε Σκυλακάκη. Έξι συνολικά έχω ζητήσει το λόγο. Και ξεκινάμε από τον κύριο Μπασίτη. Α, όχι, 7, επτά, γιατί κάλφιν έχω επίση. Επτά έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μπασίτη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μιλήσω τώρα, αφού το άκουσα και τον εκπρόσωπο του Όλαφ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένα πράγματα είναι πλέον προφανή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, Καταλίνη Βαν Σόριν. Μας έδωσε εξαιρετικές πληροφορίες και έχουμε πλέον ε, μία πλήρη εικόνα η οποία καταδεικνύει ότι στη γεωργία και στα ταμεία συνοχής εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι ήγηκε πλέον η ώρα, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, να λάβουμε μια πολιτική απόφαση εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκαν και κάποια νέα κράτη-μέλη, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, που ε, έχουν μεγάλες κλίμακας παρατυπίες. Αλλά εδώ δεν είναι, ε, πρόκειται για πολιτική απόφαση για τα κράτη-μέλη. Όταν υπάρχουν ε, εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ορθώς, θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να τηρούν τις προθεσμίες, τα χρονοδιαγράμματα και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, έχω προσωπική πείρα επί του θέματος και ξέρω πόσο στεναρά αντιστέκονται τα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν προβλήματα με τις ε, δημόσιες προμήθειες. Ε, ορισμένες φορές μπορούν να γίνουν κεντρικά τα θέματα με χρήση πληροφορικής και ελάχιστους ανθρώπους, αλλά η αντίσταση είναι πάρα πολύ στεναρή. Ε, θα περιμένω λοιπόν μια μισή ώρα για την έγκριση της Πράσινης Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να μας πούν και την άποψή τους επί του θέματος, αλλά γνωρίζω ότι ένα από τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής μας για το 2011 θα πρέπει να είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό κανονισμό για τις δημόσιες προήθειες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αίτια και όχι τις συνέπειες. Και τα αίτια αντιμετωπίζονται στα αρχικά στάδια, όταν ξεκινά μια διαδικασία. Και με το τρέχον σύστημα δημοσίων προμηθειών υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για παρατυπίες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος ε, αναφέρει ότι οι δημόσιες προμήθειες είναι το βασικό πρόβλημα. Θα πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε όλοι ότι ένα από τα βασικά μας καθήκοντα για το μέλλον είναι να έχουμε ένα διάφανο σύστημα δημοσίων προμηθειών στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον ε, φίλο Ιβάν για την έκθεσή του και να εκφράσω την ε, εκτίμηση που τρέφω για το έργο της Όλαφ. Είναι πολύ σημαντικό έργο και πιστεύω το, αναγνω... το, το καταγράφει και το αναγνωρίζει στην έκθεση του και ο εισηγητής. Άλλωστε το ακούσαμε και στις προφορικές εξηγήσει που δόθηκαν. Με δύο μόνο θέματα θα ασχοληθώ. Πρόκειται βέβαια για ένα ζήτημα περίπλοκο. Θα μπορούσα να επισέλθω στι λεπτομέρειε διαφόρων θεμάτων, αλλά δεν θα το πράξω. Το πρώτο που ακούστηκε άλλωστε νωρίτερα ήταν ε, η μέθοδος του να, και ο τρόπος του να κατανομαστούν κάποια κράτη-μέλη ή ένα κράτος μέλος. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Γιακοβέη, η οποία έχει επανειλημμένως εξηγήσει τη γνώμη της. Και έχει αναφερθεί σε στην ευρωπαϊκή ιδιόλεκτο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να κατονομάζονται οι υπέτη παρατυπιών, να δακτυλοδεικνύονται για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη ρίζα αυτών των προβλημάτων και να εξετάσουμε και τις διαστάσεις των προβλημάτων αυτών. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα ω προ τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, θα πρέπει να δούμε και την έκταση που έχει πάρει το πρόβλημα και τη ρίζα του κακού. Και βέβαια όλα τα ε, σφάλματα που έχουν παρισφρήσει στους λογαριασμούς. Χρειάζεται βέβαια πρώτα μία ε, περιγραφή των βασικών αρχών που αξιοποιούνται, που χρησιμοποιούνται στη ανάλυση. Δηλαδή να πούμε να υπάρχει διαπίστωση παρατυπιών στο τάδε και στον τάδε τομέα ε, μετά χρειάζεται ένα σαφή πίνακα που να κατονομάζει τα κράτη-μέλη. Πλην όμω, εάν δεν υπάρχουν σαφεί πληροφορίε και σαφεί αρχέ, δεν έχουμε δικαίωμα να ε, κατονομάσουμε ένα μόνο κράτο μέλος. Φυσικά εγώ δεν ε, αμφισβητώ τις καλές προθέσεις του εισηγητού και δεν καταφέρομαι κατά του συναδέλφου Ιβάν με αυτά που λέω, αλλά Έχω λίγο κουραστεί να βλέπω ε, τη χρήση επιθέτων και χαρακτηρισμών κατά καιρού που δεν στηρίζονται όμως σε πραγματικά ε, στοιχεία, σε βάσιμα στοιχεία. θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική διατύπωση. Φερρυπίν, ε, να πούμε ότι ναι, μπορεί τέτοια φαινόμενα να έχουν εμφανιστεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα μπορούσαν ενδεχομένω να έχουν εμφανιστεί και στα τάδε δίνα κράτη-μέλη και ε, το 2004 αλλά και πιο πριν ενδεχομένω, ε, πριν από την ένταξη Βουλγαρίας της Ρουμανίας, κάποιες αρχές σε κάποια κράτη-μέλη να είχαν ε, και εκείνες διαπράξει κάποιες, κάποιες φάλματα, να είχαν υποπέσει κάποιες παρατυπίες. Αλλά αυτό πάλι δεν αποτελεί λύση. Ας ξεφύγουμε λοιπόν από τον φαύλο κύκλο. Πάντα συζητούμε το πόσο ευαίσθητα αυτά τα θέματα, πάντα λέμε ε, τι δυσκολίες έχουμε από τα θέματα αυτά και ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα σαφή πίνακα των ε, παρατυπιών ε, των κρατών μελών όταν συζητούμε τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Καταλήγουμε τελικά πάντα στο ίδιο σημείο. Την αφετηρία δηλαδή το μηδέν και όπως είπε και ο εκπρόσωπος Επιτροπής πολύ σωστά δεν μπορεί να ε, κατονομάζεται ένα μόνο κράτο μέλο ή περισσότερα στη τελευταία ανάλυση, χωρί βάσιμα στοιχεία. Εγώ θέλω τώρα σαφή στοιχεία, σαφή πίνακα, με σαφεί αρχέ και ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά είναι πια το θέμα, το θέμα σοβαρό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και το ελεγκτικό συνέδριο και οι όλα έχουν επισημάνει. Υπάρχουν ε, λίγοι όμως ε, νομίζω που μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού σφάλματος. Για να λογιστείτε, αυτός ο πολίτης ε, ο οποίος ανοίγει τη σελίδα του ίντερνετ και βλέπει τον όρο ποσοστό σφάλματος δεν μπορεί να διακρίνει τι εννοεί όλο αυτό το ελεγκτικό συνέδριο με τον όρο αυτόν γιατί δεν είναι αρκετά γνώστη τη υπόθεση. Ίσα τα μία συνοχή Φερρυπίν μπορεί κανείς να δει ότι υπάρχει μείωση το ποσοστό σφάλματος αναφέρομαι στην έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου, ή να παρουσιάσετε στην έκθεση τη Όλαφ αύξηση του ποσοστού σφάλματο. δηλαδή αντιφατικά στοιχεία που παρουσιάζονται στι ιστοσελίδε στο ίντερνετ και ο πολιτή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ότι το ποσοστό σφάλματο σημαίνει άλλο πράγμα για την Όλαφ και άλλο για το Ελεκτρικό Συνέδριο. Ε, τέτοιου είδου αντιφάσεις δεν έχουμε την πολυτέλεια να παρουσιάζουμε. Uh, uh, Ευχαριστούμε κύριε Ντόιτς. Το τελευταίο που λέτε είναι σαν να συγκρίνουμε πορτοκάλια με λεμόνια. Έτσι λέμε εμείς, ότι δεν ξέρω, σε άλλες γλώσσες μπορεί να μεταφράζεται αλλιώ, λέει ο κύριος Στάς. Ο κύριος Σεντεκαρ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ για τις ε, συστάσεις που παρουσιάζονται στο σχέδιο κειμένου με τις οποίες συμφωνώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις της. Κατανοώ πολύ καλά ότι υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν θέλει να παρουσιάζει το ποσοστό της απάτης ως υπερβολικό. Αυτό το κατανοώ και το σέβομαι σε ένα βαθμό. Αφετέρου όμως δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και το πρόβλημα. όταν διαβάζω κάποια έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Θα πρέπει καταρχάς να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ απάτης και παρατυπίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ε, δεδομένο ότι πρέπει άλλο να είναι η απάτη και άλλο να είναι η παρατυπία. Αλλά όπου υπάρχουν παρατυπίες υπάρχει και ενδεχόμενο απάτης στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες τις οποίες ε, διαπιστώνονται παρατυπίες και οι παρατυπίες αυτές έκειται στο γεγονός ε, οι γεωγραφικές εκθάσεις να ε, αναφέρονται ως μεγαλύτερες από αυτές που είναι. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι υπάρχει και μια συγκεκριμένη νοοτροπία για τον τρόπο με τον οποίο μετρούνται οι συγκεκριμένε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιληφθεί ότι όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό παρατυπίας υπάρχει και ανοιχτό περιθώριο απάτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στους παραδοσιακούς ε, ίδιους πόρους και μας λέει ότι το 2009 το ποσοστό των παρατοπιών μειώθηκε. Καλά όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μου επιβεβαιώσει ότι όταν ε, εξετάζουμε τις οικονομικές επιπτώσεις ε, της ε, απάτης, έχουμε αύξηση. Υπάρχει επίσης αύξηση στις παρατυπίες για το Τομείο Συνοχής και για τη Γεωργία όπως επίσης και για τα προενταξιακά ταμεία. Και μάλιστα είχαμε αύξηση κατά αρκετές ποσοστίες μονάδες σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά λοιπόν τις άμεσες δαπάνες, ναι, έχουμε μίεση, αλλά όσον αφορά τα ποσοστά και την ονομαστική αξία σε ευρώ, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε όταν μιλάμε για απάτη, αλλά δεν μπορούμε και να υποτιμούμε το πρόβλημα και να το μειώνουμε και να το παρουσιάζουμε ως κάτι λιγότερο από ό,τι είναι. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ερώτηση τώρα. Ο εισηγητής ε, επισημαίνει το σημείο αυτό, είναι ένα θέμα όμως το οποίο προκύπτει και σε άλλες περιπτώσεις. Όσον αφορά τα προενταξιακά ταμεία για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το ΣΑΠΑΡΤ. Διαπιστώνουμε ότι η Τσεχία, η Εστονία, η Λετωνία και η Σλοβενία ε, μας ε, υπέδειξαν ποσοστά μηδέν. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ παρατυπίας για το συγκεκριμένο τομέα. Ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά. Διότι φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες. Εάν η κατάσταση είναι διαφορετική σε αυτές τις τέσσερις χώρες, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Μπορεί οι χώρες αυτές να έχουν εξαιρετική πείρα και μπορεί να γνωρίζουν πώς μπορούμε να αποφύγουμε την απάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους επόμενους να περιορίσουν λίγο το χρόνο παρέμβασής τους, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε. Επόμενος ο μιλητής είναι ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά έχω να πω. Θα περιοριστώ όμως ε, λίγα σύντομα. Για τον κύριο Ντόιτς. Ναι, θεωρητικά το naming and shaming, το να κατονομάσουμε δηλαδή τους υπετίους κάποιας παρατυπίας είναι καλή λύση, έχει αποτελέσματα, φέρνει αποτελέσματα, αλλά το πρόβλημα εμφανίζεται όταν εκείνος ο οποίος θα πρέπει να κατονομαστεί ως υπέτειος κάποιας παρατυπίας ανήκει στην πολιτική μας οικογένεια, οικογένεια και ως εκ τούτου υπάρχουν ε, ε, τα γνωστά τηλεφωνήματα από την κυβέρνηση ε, του εν λόγω κράτους, το οποίο παίρνει, η οποία παίρνει τηλέφωνο και λέει κοιτάξτε να σας πω τι γίνεται εκεί πέρα και ποιον πρόκειται να κατονομάσετε κτλ. Εκεί δυσκολευόμαστε ω προς το να κατονομάσουμε υπετήρου. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα είπε ο Σέρεν για τα τέσσερα κράτη. τα οποία παρουσιάζουν ε, μηδενικό ποσοστό απατών. Ίσως όμως καλό θα ήταν να δούμε αυτά τα κράτη και να τα ξαναπεριλάβουμε στον κατάλογο των επισκέψεών μας. Γιατί αν πάνε τα πράγματα τόσο καταπληκτικά όπως φαίνεται, καλό θα είναι να πάμε να τους επισκεφθούμε και να δούμε σε τι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Να διδαχθούμε δηλαδή από αυτή τη βέλτιστη πρακτική. Και ενδεχομένως να τους υποστηρίξουμε περισσότερο αν χρειάζεται. Και η τελευταία μου παρατήρηση. στα όσα είπε ο κύριος Πατσίτης. Είναι δυσάρεστο κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει με την έκθεση ΠΥΦ ένα κατάλογο των κρατών μελών και μετά να αποδίεται σε ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι θα συμπεριλαμβάνει αυτή η έκθεση και τελικά να πρέπει να διαπραγματευόμαστε με την Επιτροπή για το τι θα γίνει και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπό της εδώ για τα όσα είπε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όταν συζητούμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ιδιαίτερα σε επίπεδο επιτροπή προπολογισμών, ίσω υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα πίεση σε σχέση με το Συμβούλιο. Και εκεί ίσω μπορούμε να περιμένουμε ότι και στις προσεχείς διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα έχουμε αντίστοιχες, ε, αντίστοιχο γλέντι όπως ε, και πέρυσι. Εν πάση περιπτώσει την έκθεση ΠΙΦ θα πρέπει να τη δούμε ιδιαίτερα στις λεπτομέρειες που αφορούν τα κράτη-μέλη στα οποία παρουσιάζονται κάποια προβλήματα και να ε, υποβάλουμε αυτά τα θέματα για συζήτηση στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ ότι για παραδείγματα χωρών, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ζητήσουμε έναν κατάλογο με όλες τις χώρες και με όλα τα ποσά, με όλα τα νούμερα. Έτσι πρέπει να δουλέψουμε. Αυτή είναι η αποστολή μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να δούμε τι κάνει κάθε χώρα μέλος. Και να δούμε τα νούμερα για όλες τις χώρες, είτε πρόκειται για παρατυπίες, είτε για πάτες κλπ. κλπ. Θέλω να πω ότι και η Όλαφ και η Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο το ίδιο πρέπει να κάνουν. Και αν θέλουμε μια πολιτική και μια στρατηγική για το μέλλον, πρέπει να έχουμε τα νούμερα για όλες τις χώρες μέλη κάθε μία ξεχωριστά. Τώρα, δύο λόγια για την έκθεση. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή. Πολύ σύντομα, θέλω να σας πω ότι κοιτάω το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών και εδώ θα ήθελα μία λεπτομερή μεθοδολογία για το νέο αυτό σύστημα διαχείρισης παρατυπιών θα ήθελα πληροφορίες ήδη από φέτος για το τι θα γίνει του χρόνου. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τον αριθμό των παρατυπιών που έχουν αναφερθεί βάσει του νέου αυτού συστήματος διαχείρισης παρατυπιών. Και το λέω γιατί άλλες μεθόδους χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη και αλλιώς εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί, ελπίζουμε, το νέο σύστημα και ίσως έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Κάτι επίσης που με ανησυχεί, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι ότι μερικές χώρες αναφέρουν πολύ χαμηλά επίπεδα παρατυπιών. Ιδιαίτερα εκεί όπου η χρηματική ενίσχυση είναι ιδιαίτερα υψηλή. Θα ήθελα επίσης να ασχοληθούμε με το θέμα των παρατυπιών και των απατών διαφορετικά στην κάθε περίπτωση. Οι απάτες σε σχέση με τις παρατυπίες στον τομέα των ιδίων πόρων είναι κάτι που με απασχολεί πολύ για μερικές χώρες επίσης ότι οι απάτες είναι πάνω από το μισό του ποσού σε κάθε χώρα μέλος. Υπάρχουν επίσης πολλές παρατυπίες ή δηλώσεις για μη εισπραγμένα ποσά και δεν ξέρω, τώρα θέλω να αρχίσω καινούργια συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να αναφέρονται ή όχι ε, με το όνομα κάθε φορά και έπειτα να δούμε και τη σύνδεση της διαφθοράς με τις απάτες. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μακαβέ. Δεν ήξερα ότι ήσασταν σκιώδη εισηγήτρια. Αλλιώς θα σας είχα δώσει το λόγο νωρίτερα, ε, συγγνώμη. Ο κύριος Κυλακάκης τώρα. Thank you, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον συνάδελφο για τη τόσο καλή δουλειά που έχει κάνει. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και αυτό είναι η μέτρηση της απάτης και της διαφθοράς. Η Επιτροπή λέει και τους έχουμε ακούσει ότι δεν μπορεί να το κάνει, δεν γίνεται. Είναι αλήθεια ότι τα μέσα που έχουμε στη θέση μα μέχρι τώρα δεν φτάνουν και είναι αλήθεια επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει αυτά έτσι τα συστήματα που δεν είναι τόσο λεπτομερή, εκτός συνόρων μας, στην αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την διαφάνεια. Είναι ένας τρόπος για να ασχοληθούμε με τις χώρες όπου η διαφθορά είναι πάρα πολύ ψηλή. Τώρα η μέτρηση της διαφθοράς είναι κάτι με το οποίο επιστημονικά έχω ασχοληθεί. Κοίταξα λοιπόν λίγο τι έχει γραφτεί, τι λένε τα διάφορα επιστημονικά δοκίμια σχετικά και που είναι όλο και περισσότερα την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν νέα πράγματα που συμβαίνουν. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ερευνήσουμε και να δούμε τι επιστημονικοί τρόποι υπάρχουν για να μετρηθεί η διαφθορά και η απάτη πέρα από την συνήθεια διαδικασία που ακολουθούμε εδώ και που είναι να μετράμε ή τη διαφορά ή την απάτη. Ρίχνουμε το δίχτυ και ό,τι πιάσουμε. Αν έχει μεγάλα μάτια θα πιάσουμε λίγα. Αν το δίχτυ έχει μικρά μάτια θα πιάσουμε περισσότερα ψάρια. Να δούμε μήπως υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέτρησης όμως. Ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει για μικρής κλίμακας διαφθορά, έτσι ονομάζεται τουλάχιστον, στη γλώσσα του τομέα, που είναι πολύ σημαντικό στη γεωργία. Γιατί στη γεωργία υπάρχουν τρόποι να μετρηθεί η διαφθορά ακόμα και με δημοσκοπήσεις. Αν μιλάμε τώρα για μεγάλη κλίμακα διαφθορά, εκεί χρειαζόμαστε διαφορετικού τρόπου μέτρηση φυσικά. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω δει τίποτα στα ερευνητικά προγράμματα για τη μέτρηση τη διαφθορά. Αν πούμε απλώ, Α, δεν μπορούμε, δεν γίνεται, και δεν κάνουμε τίποτα, καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια, δεν θα γίνει και ποτέ. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι καινούριο βγαίνει, τι μέθοδοι υπάρχουν και εμείς πρέπει να το προωθήσουμε αυτό. Γιατί αν δεν μπορούμε να μετρήσουμε, τότε δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν ξέρουμε αν τελικά πιάνουμε τα μικρά ή τα μεγάλα ψάρια. Δεν ξέρουμε αν είμαστε αποτελεσματικοί ή απλώς ε, καθόμαστε και κοιτάμε. Είμαστε κομπάρσι σε όλη αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε κύριε Σκυλακάκη. Νομίζω ότι σωστά τα λέτε. Αλλά εδώ δεν σας βλέπω καλά. Από ό,τι όμως βλέπω, όπως κινούνται αυτοί οι εκπρόσωποι της Επιτροπής εδώ πέρα, τους βλέπω ότι θέλουν να αντιδράσουν σε αυτά που είπατε. Κάτι θα έχουν να πούνε. Έχω την εντύπωση ότι ναι, κάτι θα έχουν να πούνε. Ο κύριος Σκάλφιν τώρα. Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο δεν είναι σχετικό με τα όσα συζητούμε τώρα. Γιατί οι περισσότεροι είμαστε και μέλη της Επιτροπής των Προπολογισμών και θέλω να επισημάνω ότι συχνά συμπίπτουν οι συνεδριάσεις των δύο επιτροπών και κυρίως οι ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν στο μέλλον να αποφεύγουμε τέτοιου είδους επικάλυψη. Δεν μπορούμε να κινόμαστε πανταχού παρόντες. Για την έκθεση λοιπόν. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ τον εισηγητή. Η έκθεσή του είναι στο σωστό δρόμο και πιστεύω ότι η Επιτροπή του Ελέγχου των Προϋπολογισμών έχει χάρη στην έκθεση αυτήν ε, ένα μηχανισμό χάρη στον οποίο μπορεί να εξασφαλίσει την καταπολέμηση κάθε μορφή απάτης και κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βεβαίω, όταν έχουμε στοιχεία είναι εύκολο να τα συγκρίνουμε. Οι αναλύσει όμως θα πρέπει να γίνονται με πολύ προσεκτικό τρόπο. Γιατί εύκολα πέφτει κανείς στο σφάλμα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα που αφορά τη χώρα μου. Το 2008, κατόπιν ελέγχων που επέβαλαν η Επιτροπή και η Όλαφ, ήρθε η καταβολή των πληρωμών, μια από τις πιο σοβαρές ποινές που μπορεί να επιβληθεί σε μια χώρα. Και αυτή η άρση αποτελεί καλό παράδειγμα των πρακτικών που ακολουθεί η Επιτροπή και η Όλαφ. Ύστερα από την λήψη από πλευρά της χώρας με μέτρων ε, ε, έγιναν οι έλεγχοι το 2009 και στη συνέχεια ξεκίνησαν και πάλι οι πληρωμές. Όμως στην έκθεση δίνεται ένα στοιχείο που έχει αναφέρει, που προθέτεται απορρέει από την βολγαρική κυβέρνηση για 20% ποσοστό ε, παρατυπιών, ε, απατών, ε, και καταβληθεί των ποσών. Και αυτό βέβαια είναι πολύ επώδυνο να το βλέπει κανεί όταν σε άλλε χώρε το αντίστοιχο ποσοστό είναι 1%. Εν πάση περιπτώσει, ε, ήρθε όπω είπα το σύνολο των πληρωμών και μετά όταν διορθώθηκαν τα προβλήματα επαναλήφθηκαν οι πληρωμέ. Ίσως υπάρχει τρόπος να εξηγηθεί το πρόβλημα διότι φαίνεται ότι ε, απεστάλει κάθε σχέδιο που είχε υποβληθεί για χρηματοδότηση στην ε, εισαγγελία, δηλαδή, και πιστεύω θα με στηρίξουν σε αυτό που λέω οι συνάδελφοι, ε, το πρόβλημα, μάλλον τα ποσοστά εξηγούνται από το ότι ήταν πολύ, ότι δεν έγινε καμία διάκριση μεταξύ παρατυπίας ή απάτης. Αυτό έχει όμως πολύ σημαντικές συνέπειες διότι φτάσαμε μέχρι χρεοκοπίας πολλών ε, επιχειρήσεων που αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν μπορούσαν να λαμβάνουν σχέδια προς εκτέλεση. Άρα, έχουμε ένα ζήτημα με τις στατιστικές, έχουμε ένα ζήτημα με τους ελέγχους που ε, γίνονται εξ εκ των υστέρων, έχουμε ένα πρόβλημα με προτεραιότητες που δεν είχαν προσδιοριστεί ικανοποιητικά. Εν τω μεταξύ, βέβαια, η σχετική υπηρεσία ε, διόρθωσε τον τρόπο λειτουργίας της και έτσι ίσως κερδίζονται κάπως αυτές οι μεγάλες διαφορές. Για να επανέλθω λοιπόν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, όταν μιλάμε με νούμερα, τα νούμερα πρέπει να στηρίζονται σε μια καλή, σωστή ε, και πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η Όλαφ να θεσπίσει μια μεθοδολογία που θα μας επιτρέπει να έχουμε συγκρίσιμα αριθματικά στοιχεία. Επίσης άλλο ένα παράδειγμα από το 2004, 88,5% των απατών εισφαλμάτων στις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Είναι δυνατόν αυτό. Κάπου πρέπει να υπάρχει λάθο. Δεν μπορεί 9 στα 10 σχέδια που έχει να λάβει μια, μια επιχείρηση ή επιχειρήσει σε μια χώρα που κατά τα άλλα έχει καλέ επιδόσει να είναι ε, λάθος, να είναι αντικείμενο κακοδιαχείρισης και απατών. Εάν λοιπόν θέλουμε και να προβάλλουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιπερασπιστούμε και να καταπολεμήσουμε τι απάτε, πρέπει να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Ευχαριστούμε. Η παρατήρησή σας έχει να κάνει βέβαια και με την Επιτροπή Προεπολογισμών. Εμείς έχουμε κοιτάξει ότι δεν συμβαίνει συχνά οι δύο γραμματείες να προσπαθούν να συντονίζονται. Η μόνη στιγμή που θα μπορούσε να συμβεί είναι 3 Μαρτίου να έχουμε κοινή συνάντηση. 3 Μαρτίου που συνεδριάζουμε εμείς και στην Επιτροπή Προπολογισμών προβλέπεται, αλλά με επιβεβαίωση ακόμα, μια συνεδρίαση. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συνεδρίασή του στις 3 Μαρτίου, μπορούμε μαζί να συναντηθούμε με την Επιτροπή Προπολογισμών. Η κυρία Ιβάνοβα είναι η τελευταία. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα διάφορα προβλήματα, οπότε εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και να κάνω και μια έκκληση. Όταν κάνουμε αξιολογήσεις, όταν κάνουμε συστάσεις, να είμαστε αντικειμενικοί. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής το έχουν προσθέσει, έχουν επιμείνει στο ότι ο κατάλογος των χωρών θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πλήρης, πιο μεγάλος. Αν υπάρχει απάτη, αν υπάρχει σφάλμα, πρέπει να υπάρχει σε ένα κατάλογο που να είναι πιο πλήρης από αυτόν που έχουμε τώρα. Να μην καταδεικνύουμε μία μόνο χώρα για κάτι το οποίο μπορεί να έχει συμβεί πριν από μερικά χρόνια. Όσον αφορά την Βουλγαρία, ναι, φυσικά έχουν γίνει αλλαγές ε, τα είπε και ο συνάδελφος. Οι πληρωμές σταμάτησαν το 2008, αλλά στη συνέχεια, μετά από τα μέτρα που υιοθέτησε η βουλγαρική κυβέρνηση, οι πληρωμές άρχισαν και πάλι να γίνονται. Άρα να είμαστε αντικειμενικοί μην τα βάζουμε με μια χώρα, να είμαστε αντικειμενικοί παρακαλώ και να κάνουμε μια καλή σύγκριση επί ίσης όρης και βάσει των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από τις διάφορες χώρες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής τώρα παρακαλώ να απαντήσουν στις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν. Αναφέρθηκαν διάφορα για το ψάρεμα, την αλία. Τι ψάρια ψαρεύουμε, ακούσαμε. Ποιος θα απαντήσει από εσά. Παρακαλώ, ποιος θέλει, παρακαλώ. Ξεκινήστε, δεν είναι απαραίτητο να είναι ο κύριος Ιλέτ, ποιος θέλει εσείς. Παρακαλώ κύριε Ιλέτ. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκπρόσωπος από κάποια άλλη γενική διεύθυνση που να θέλει να λάβει το λόγο. Αν όχι κύριε Πρόεδρε, θα αναλάβω εγώ την ευθύνη και θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Όλαφ ταυτοχρόνως. Ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, κάποιες ιδιαίτερως τεχνικές και δεν θα κάνω καμία απόπειρα να απαντήσω σε όλες εδώ. επανέρχεται συνεχώς το θέμα της διαφοράς μεταξύ απάτης και παρατυπίας, διότι η απάτη είναι παράτυπη, αλλά δεν είναι όλες οι παρατυπίες απάτη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσω το ίδιο θέμα, απλώς να πω ότι θα πρέπει από τα στοιχεία που έχουμε για τις παρατυπίες θα πρέπει να εμβαθύνουμε για να διαπιστώσουμε ποια είναι η στοιχεία απάτης αν ε, πάρω το παράδειγμα της, ε, ε, των υπερβολικών δηλώσεων μεγαλύτερων εκτάσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι αποτέλεσμα αποφάσεων των γεωργών για να δηλώσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση η όλα θα πρέπει, θεωρεί ότι θα πρέπει να το εξετάσουν οι εθνικές αρχές για να δούνε αν ε, υπάρχει απάτη στην κάθε δήλωση και αν υπάρχει και θέμα το οποίο είναι ενδιαφέροντος ε, του κράτους μέλους. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι όταν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπήρχε στατιστικά υπερβολική δήλωση θα περάσει σε δημοσιονομική διόρθωση που βάσει του συστήματος θα χτυπήσει τον εθνικό προπολογισμό και θα υπάρχουν συνέπειε εκεί. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα του τι προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις και με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τομείς. Τώρα για το πολύ δύσκολο θέμα για τις ε, μελέτες, για τις ε, διορθώσεις, ε, ούτε ήθελα να μιλήσω, δεν το έχω κατανοήσει ούτε κι εγώ ακόμα αρκετά καλά και ελπίζω ότι θα έχουμε χρόνο όταν θα έρθει ο νέος Γενικός Διευθυντής και νομίζω ότι θα καθίσουμε κάτω με τον Διευθυντή και θα ασχοληθούμε με το θέμα, το ελπίζω τουλάχιστον. Ο κύριος Κυλακάκης έχει δίκιο από ενοιολογικής πλευράς. Θα πρέπει να το εξετάσουμε καθημερινικώς, πέρα από το πλαίσιο και τους περιορισμούς που προκύπτουν όταν ε, εφαρμόζουμε τη δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει να το δούμε και εκτός αυτού του πλαισίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ετοιμάσει και μια στρατηγική κατά της διαφθοράς και μια στρατηγική κατά της απάτης. Τα δύο έγγραφα αυτά θα είναι έτοιμα στη διάρκεια του έτους και θα λάβουμε υπόψη και τα όσα έχουμε ακούσει κατά την προετοιμασία τους. Για τις τέσσερις χώρες οι οποίες αναφέρονται ε, με μηδενικό ποσοστό παρατυπιών, θα πρέπει να σας πω ότι οι επιθεωρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάτι λανθασμένο στα όσα δήλωσαν. Δεν έχουν διαπιστωθεί πολύ σημαντικά λάθη στα προγράμματα αυτά, στις χώρες αυτές, στους ελέγχους που έγιναν. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση την οποία θα έπρεπε να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις διάφορες παρατηρήσεις. Ο κύριος Ιβάν πρέπει να φύγει και άρα δεν μπορεί να αντιδράσει. Νομίζω ότι ήταν επικοδομητική η συζήτηση που είχαμε με πολλές παρατηρήσεις. Ακούστηκαν και μερικές διαφορές μεταξύ μας. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο τώρα ώστε να τροποποιηθεί η έκθεση ΒΑΝ μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Τότε λύγει η πρόθεση για την, για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε την έκθεση ΒΑΝ στις 28 Φεβρουαρίου υπό την Προεδρία Ντεματζίστρης ελπίζω και στην Ολομέλεια προβλέπεται να συζητηθεί στην μήνυ Ολομέλεια 23 και 24 Μαρτίου εδώ στις Βρυξέλλες. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο 4. Εδώ έχουμε κάποιους προσκεκλημένους από την Deloitte. Είναι εδώ. Έχουν ετοιμάσει το έγγραφο το οποίο έχουμε και εμείς μπροστά μας. Έχει μοιραστεί, είδα από την προηγούμενη εβδομάδα, φαντάζομαι το έχετε μαζί σας. Είναι ένα ενδιαφέρον έγγραφο για ένα θέμα που είναι συναρπαστικό πιστεύω. Γιατί υπάρχουν νέα σημεία στη συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά αυτό το θέμα. Από ό,τι κατάλαβα έχετε και μια παρουσίαση PowerPoint, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Λέγομαι Φρανκ Στάλενς, είμαι εδώ με τον συνάδελφο Ρίτσαρντ Όχερστη. Είμαστε και οι δύο ε, μέλη της Deloitte. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης μελέτης ε, του Ευρωπαίου, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταρχάς, να κατανοήσουμε το στόχο της μελέτης. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν ε, να δούμε σε τι σημείο βρίσκονται οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην, ε, στο ποινικό δίκαιο και την προστασία των ε, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά σε σχέση και με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Από αυτό το πρίσμα λοιπόν αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών. Καταρχάς ε, τις απαντήσεις, ερωτολόγια και συνεντεύξεις από τους εκπροσώπους των διαφόρων οργανισμών, τη Eurojust, ε, τη Europol και την Olaf. Επιπλέον, λάβαμε και κάποια στοιχεία από όσους συμμετείχαν στα πρόσφατα σεμινάρια επί του θέματος και έγινε και έρευνα ε, για τις ε, πηγές ε, δημοσίων αναφορών. Να περάσουμε απευθείας λοιπόν στα βασικέ βασικές μας διαπιστώσεις. Καταρχάς, φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανισμών. Κατά τα φαινόμενα υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας, αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχει το πλαίσιο συνεργασίας, η ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται εντό των ε, συμφωνιών συνεργασίας δεν φαίνεται να εφαρμόζεται πλήρως στην πράξη. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η συζήτηση είναι πολύ δραστήρια, το θέμα είναι ε, επίκαιρο και υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις από τους ενδιαφορομένους για την προστιθέμενη αξία του EPPO, του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, και την ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο γραφείο. Βάσει των τριών οργανισμών υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση αντικτύπου και αξιολόγηση των αναγκών. Επίσης αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο είναι περαιτέρω προκειμένου να δοθούν ε, απαντήσεις σε πιο διεξοδικές ερωτήσεις ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει μια αναδιοργόνωση σε περίπτωση που δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θεωρείται ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να προετοιμαστούμε για μελλοντικές αποφάσεις. Και οι τρεις οργανισμοί επίσης ε, συμφωνούν για την ε, προστιθέμενη αξία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και με ανεξάρτητη ε, δυνατότητα ποινική έρευνας και ανάκρισης και επίσης προσπαθούν να έχουν ένα ισότιμο επίπεδο προστασίας στα κράτη-μέλη και πιστεύουν ότι με αυτό θα επιτευχθεί. Και οι τρεις επίσης συμφωνούν ότι είναι λογικό για τις εξουσίες που δίνονται για έρευνα για σοβαρά εγκλήματα τα οποία δια, ε, διαπράττονται από, από υπαλλήλου των ευρωπαϊκών οργάνων αυτά να πηγαίνουν σε κάποιο ανώτερο δικαστικό σώμα. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα Βάσει των στοιχείων που μας έδωσε η Όλαφ, ε, φαίνεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε συνένεση ε, και να είναι η Eurojust ε, το ανεξάρτητο όργανο για τη, που θα δράσει στα αγγελία στα κράτη-μέλα, ενώ η Europol και η Όλαφ θα μπορούν να κάνουν τις έρευνες και τις ανακρίσεις για τους ε, Ευρωπαίους ανακριτές. Επίσης, η Όλαφ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό συμβουλευτικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα δίνει συμβουλές στους ε, ανακριτές της Όλαφ και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν και γραφεία εισαγγελίας, και θα υπάρχει ανεξάρτητη δράση μόνο όταν τα, οι αρχές των κρατών μελών δεν μπορούν να δράσουν. Η Όλαφ επιπλέον θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι ανακριτές θα πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της Europol για να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ε, στις έρευνες και τις ανακρίσεις που γίνονται. Όπως σας ανέφερα την αρχή της παρέμβασής μου, συμμετείχαμε σε όλα τα πρόσφατα σεμινάρια επί του θέματος. Ε, το στρατηγικό σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο πέρσι από τη Eurojust σε συνεργασία με τη Βελγική Προεδρία καθώς επίσης και το ετήσιο φόρουμ για την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων ε, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τον Οκτώβριο. Στα σεμινάρια αυτά λάβαμε και κάποιες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες και από τα στοιχεία που λάβαμε από αυτούς θεωρείται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Eurojust. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει και βάσει των συμμετοχόντων υπάρχουν και οργανωτικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ε, υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια για τη σχέση μεταξύ των δύο και τα σενάρια αυτά είναι τα εξής. Η Eurojust να γίνει μια ευρωπαϊκή εισαγγελία με σταδιακή αύξηση των εξουσιών της ε, και χώριση εξουσιών από τα κράτη-μέλη ή η Ευρωπαϊκή Συγγελία δρά ω ανεξάρτητο φορέα από κοινού με τη Eurojust και τους υπολείπου. Ε, δημιουργείται ένα ειδικό τμήμα στη Eurojust Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ένα τελευταίο σενάριο. Συγχωνεύονται τα δύο για να αποτελούν έναν φορέα αλλά με διαφορετικές δομές λήψης αποφάσεων. Στη διάρκεια του ετήσιου φόρου λάβαμε και κάποια στοιχεία από τους εθνικούς δικαστές και εισαγγελείς αυτοί θα προτιμούσαν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μια παράλληλη προσέγγιση η οποία θα ενισχύει ταυτόχρονα τη Eurojust αλλά θα ε, αναπτύσσει και περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι βασικές μας συστάσεις τώρα καταρχάς η άποψή μας είναι ότι είναι πρόημο αυτή τη στιγμή να δώσουμε ενδελεχείς συστάσεις ιδίω για περίπλοκα θέματα όπως είναι η αρχιτεκτονική θεσμική δομή της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Και τούτο διότι ερίζουν οι απόψεις επί του θέματος. Ε, επίσης δεν είναι σαφές το θέμα στη συνθήκη και υπάρχει και διαφωνία για ε, τα πιο ουσιαστικά ε, θέματα μεταξύ των διαφέρων οργανισμών και επίσης όπως σας είπα και στην αρχή το γεγονός ότι οι διάφοροι οργανισμοί είναι διατεθειμένοι να δώσουν πιο ενδελεχείς απαντήσεις μόνο εάν ε, γίνει αξιολόγηση αντικτύπου και αξιολόγηση των περαιτέρω αναγκών. Όμως είμαστε προετοιμασμένοι να φροντίσουμε την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών, να κάνουμε περαιτέρω ε, αξιολογήσεις αντικτύπου και αναγκών και να διοργανώσουμε και πιο διαρθρωμένες συζητήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων και των αρχών των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κάνει μία σύσταση προκειμένου να ενισχύει η Eurojust και να δούμε πώς μπορούμε να ε, προτείνουμε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να έχουμε μια πιο ενημερωμένη άποψη του, του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε η Επιτροπή. μήπω υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, ο οποίος θέλει κάτι να πει για την κατάσταση πραγμάτων. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής εισαγγελία ή σε σχέση με αυτά που μας προτείνει η Deloitte. Συγκρίνοντάς τα με αυτά που σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάποιος εδώ. Εγώ είχα καταλάβει ότι υπήρχε κάποιο, ο κύριος Μισελίνη, από την Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη. Ή όχι. Εσείς είστε ο κύριος Μισελίνη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ χαιρόμαστε για την μελέτη αυτή είναι ευπρόσδεκτη, είναι πολύ χρήσιμη. Παρουσιάζει την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα με σαφήνεια. Και επίσης αντικατοπτρίζει κάπως και την ιστορία της Eurojust, Europol και μιλάει για την ιδέα αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επιβεβαιώνουμε και εμείς ότι πράγματι ε, δουλεύουμε πάνω στις θεσμικές δυνατότητες που υπάρχουν ώστε βάσει του άρθρου 85 και 86 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως μπορούμε να προχωρήσουμε. τίθεται θέματα νομικά, λειτουργικά, τα οποία πρέπει να μελετηθούν σε βάθος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως και οι υπηρεσίες της το μελετούν όντως σε βάθος και ζητάμε και την συμμετοχή όλων των διαφερομένων και των κρατών μελών προκειμένου να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε από την πλευρά της μία μελέτη για την ενίσχυση της Eurojust. Γίνεται κατά τη διάρκεια του 2011. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη της χρονιάς. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει και ανακοίνωση για τη δυνατότητα δημιουργίας ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2013. Έχει προχωρήσει σε διαβούλευση και μελέτη. Αυτή είναι η κατάσταση πραγμάτων. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο και επαναλαμβάνω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την μελέτη που μόλις παρουσιάστηκε. Πρόεδρος, η κυρία Γιάννα Σέντερ έχει ζητήσει το λόγο μόνο για αυτό το θέμα. Άλλος κανείς? Σέντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη και για την παρουσίαση που ακούσαμε. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ και καλό θα ήταν να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμείς κάποια πρόταση για την εισαγγελία αυτή. Θέλω να ρωτήσω κάτι τους ειδικούς. Πρώτον, Από αυτά που ακούσαμε φαίνεται ότι η διαβούλευση, σεμινάρια κτλ. δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει συνένεση υπέρ του ότι η Eurojust να είναι πώς το πω, η έδρα της εισαγγελία και να αποτελείται από δύο σκέλη, τη Europol και την Olaf που θα ερευνούν, θα κάνουν την αστυνομική δουλειά. Τώρα εσείς που είσαστε ειδικοί, γιατί άλλο τι λένε οι άλλοι, εσείς που είσαστε ειδικοί, βλέπετε όντω να υπάρχει τέτοια συνένεση και από πλευρά ελέγχου προπολογισμού μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτά τα δύο σκέλη, για να τα πω έτσι, που θα βοηθάνε την Eurojust, η αυτά δηλαδή και η Europol. πώς θα είχαν οι δραστηριότητες, ε, τι τύπου θα ήταν, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, ποια είναι τα δυνατά και οι αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και αδυναμίες από ένα τέτοιο σύστημα με δύο ανακριτικές αρχές. Η ξέρουμε ότι ιστορικά ερευνά τις απάτες στην Επιτροπή Άρα εντάσσεται μέσα στην Επιτροπή. Τώρα με το νέο αυτό σχήμα θα έβγαινε οριστικά η Όλαφ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε πώς το βλέπετε αυτό. Έπειτα μιλήσατε για επικαλύψεις. Είναι όντως ένα από τα προβλήματα που μας απασχολούν και μας πολύ. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι επικαλύψεις υπάρχουν. Ποιες είναι οι επικαλύψεις που θα έπρεπε να αποφύγουμε. Έπειτα, εισαγγελίε των χωρών μελών και οι δικαστικές υπηρεσίες δεν είναι και πολύ υπέρ μιας ευρωπαϊκής εισαγγελία. Λένε ότι καλύτερη είναι η συνεργασία για αυτούς. Και για τη Eurojust το ίδιο ισχύει. Γιατί οι χώρες μέλη συμμετέχουν στη Eurojust κανονικά. Αλλά ποια είναι η άποψή τους, όπως ξέρετε. Και κάτι ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει, όταν δεν διαπιστώνεται σαφήνεια στις συνθήκες από τους ειδικού Πώς θα μπορούσαμε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά όπου λείπει η σαφήνεια για τα άρθρα 85-86 κάπου αλλού στη συνθήκη. Ε, μπορεί να γίνει κάτι για να αποσαφινιστούν αυτά τα σημεία και να προχωρήσει η διαδικασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Άλλος κανένας συνάδελφος παρακαλώ που έχει ερωτήσεις. Από την Deloitte τίποτα. Καλά, τότε να απαντήσει η Deloitte. Ποιος θα απαντήσει, ένας από τους δύο αποφασίστε ποιος θα μας απαντήσει. Παρακαλώ, κύριος Ντάλλας. Of Σαφώς και μπορούμε να απαντήσουμε, παρά το γεγονός ότι θέσετε πολλές ερωτήσεις. Um, as ε, Όπως αναφέρατε επίσης, ακόμα πλέουμε σε βαθιά νερά και δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες για επικαλύψεις και την καλύτερη άγουσα που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Θα πρέπει να γίνουν εις βάθος συζητήσεις με τους διάφορους οργανισμούς. Όταν ε, έθεσα τα ερωτήματα για το πού διαπιστώνουν ότι θα υπήρχε αλληλεοπικάλυψη μεταξύ τους, ε, η απάντηση ήταν, όπως σας είπα και προηγουμένως, χρειάζεται μεγαλύτερη αξιολόγηση αντικτύπου για να μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Επίσης, να σας πω ότι όταν έστειλα τις απαντήσεις από τους διάφορους οργανισμούς, ε, από τον ένα στον άλλον, ο καθένας τους απάντησε ότι ήταν πολύ νωρίς για να απαντήσουν για τις απαντήσεις από τις άλλους ε, οργανισμούς γραπτός. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να διοργανηθούν ε, συνεδριάσεις για να γίνουν πιο διαρθρωμένε και ει βάθο συζητήσει μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Πέραν αυτού βέβαια, Δεν ξέρω αν έχετε και κάτι άλλο, γιατί ειλικρινά σας ομολογώ ότι το ξέχασα το μεγαλύτερο τμήμα των ερωτήσεών σας. Τότε ευχαρίστω να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ για να επαναλάβει. Ναι, παρακαλώ. Ε, ναι. Με ανησυχεί λίγο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι μελέτες. Δηλαδή, όταν αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο θεωρώντας ε, ότι για ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα στα σπάργανα, αν θέλετε, το να στέλνουμε λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο σε αυτούς ε, οι οποίοι πρέπει να καθορίσουν, να απαντήσουν ε, αν η θέση μου είναι θετική ή αρνητική, είναι λίγο ασαφές. Θα έπρεπε να αναλύσουμε λίγο καλύτερα ε, τι στάση έχουν, ε, τι σχέσεις έχουμε μαζί τους, γιατί το να τους στέλνουμε ένα ξερό ερωτηματολόγιο ε, δεν είναι τρόπος να κάνουμε τη μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι εκ των προτέρων ότι θα λάβουμε ελάχιστες απαντήσεις. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι συγκεκριμένα. Ε, θα έπρεπε να δούμε λίγο και τι γίνεται με την εμπειρία μας, ε, τι έχουμε να πούμε από τις εκθέσεις που κάνουμε. Στις συζητήσεις μπορεί να υπήρχαν προβλήματα με τη Γιούλοφ, με τη Europol, ε, να ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται. Το να του στέλνουμε ένα ερωτηματολόγιο έτσι σκέτο ήταν πολύ δύσκολο να μας οδηγήσει σε καλές απαντήσεις. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας ρωτήσω είναι και σας ευχαριστώ γιατί φαίνεται να έχουμε μια καλή τάση. Ε, από όλε λοιπόν τις απαντήσεις που λάβαμε, φαίνεται να υπάρχει μια κάποια συνένεση. Να είναι δηλαδή η Eurojust η έδρα αν θέλετε, αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ω εισαγγελία που φαίνεται και το πιο λογικό και από εκεί και πέρα να έχει και δύο διακλαδώσει την Όλαφ και την Europol. Αν έχουμε λοιπόν ε, ε, κάποιον στην κεφαλή και δύο ε, άκρα από την δεξιόν και εξ αριστερών, ποιος θα είναι ο ρόλος της Όλαφ σε αυτή τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων ιστορικώς υπάρχει το εξής πρόβλημα με την Όλαφ. Οι αρμοδιότητες τους είναι η καταπολέμηση της απάτης Εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια υπηρεσία η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή μου είναι, σε αυτό το τρίγωνο λοιπόν που έχουμε, τη Eurojust, τη Europol και την Olaf, η Olaf θα συνεχίσει να είναι τμήμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία που θα εξαρτάται περισσότερο από τη Eurojust, αλλά φυσικά θα την πληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, λέτε σαφώ ότι δεν είναι αρκετά σαφή η συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι εξετάζει τι γίνεται με τα άρθρα 138 και 136. Θα ήθελα να μου πείτε όταν μιλάτε για ασάφεια ε, σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Ποια είναι τα σημεία που δεν είναι σαφή. Τελευταία ερώτηση. Στην ε, τελευταία διάσκεψη εισαγγελέων και δικαστικών ε, ευρωπαϊκών σωμάτων φαίνεται ότι υπήρχε γενικότερη άποψη να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να μην υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινοτικό σώμα εισαγγελία. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για τη σχέση μεταξύ αυτών των ε, ε, εισαγγελιών των 27 κρατών μελών και της Eurojust, διότι μια κάποια συνεργασία υπάρχει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία για να φτάσουμε σε ένα στάδιο παραπάνω από τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θεωρώ ότι προσθέμενη αξία προσφέρει αυτή η μελέτη έγκυται στο γεγονός ότι κάθε ενεργό σώμα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την γνώμη του, τη θέση του σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και επίσης καθιστά σαφές ότι τα διάφορα σώματα, όργανα πρέπει να συνεργαστούν το ταχύτερο δυνατό και να προβούν σε εις βάθος συνομιλίες. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι πέραν των ερωτηματολογίων οργανώνουμε και συνεντεύξεις. Άρα έχουμε συνεντεύξεις με ενώπιος ενωπίων επικοινωνία με τον κάθε φορέα από αυτούς. Πέραν των γραπτών απαντήσεων που έχουμε λάβει. Ως ανεξάρτητη αρχή λοιπόν, και ανέφερα νωρίτερα ότι είμαστε ανεξάρτητη αρχή, οργάνωση που παράγει ανεξάρτητη μελέτη. Εάν διαπιστώσουμε σημαντικές διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ κυρίων παραγόντων της διαδικασίας αυτής και ιδιαίτερως ως προς το ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν, ασφαλώς ως ανεξάρτητη αρχή δεν είμαστε θέση να λάβουμε εμείς την απόφαση για λογαριασμό του. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε τις διαφορές, τις αποκλήσει απόψεων που υφίστανται. Και ήδη ανέφερα νωρίτερα ότι πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των αναγκών, μια πρόβλεψη του τι θα χρειαστεί στο μέλλον και πώς θα πρέπει να οργανωθεί το τι θα προβλεφθεί και πώς θα συνεχίσουν αυτοί, αυτές οι αυτοί οι παράγοντες να εργάζονται. Και ταυτόχρονα βελτιώσεις που παραλαμβάνω δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια, αλλά προφορικά από τις συμμετοχές στο σεμινάριο βλέπουμε διαφορετικές επιλογές για την ε, νέα οργάνωση, για μια νέα οργάνωση της Όλαφ. Μία από τι προτάσει που ακούστηκε στο σεμινάριο ήταν να ε, τριχοτομηθεί η Όλαφ, να υπάρχει μια διοικητική δομή, μια εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου που θα υπαχθεί στο ελεκτικό συνέδριο και μια ε, πάταξη των απατών που θα υπαγόταν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση και διάλογος μεταξύ των διαφορών όπως παφορέων και ε, θεσμικών οργάνων. Αυτό για να μπορούμε να έχουμε και καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Για αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνένεση για το ποιο είναι το ερευνητικό σώμα, ποια είναι η διοκτική αρχή. Όλαφ, Europol και οι δύο θεωρούν ότι έχουν ρόλο διοκτικό. Όσον αφορά την ε, ασάφεια σε επίπεδο διατύπωση συνθήκη, υπάρχουν νομίζω διαφορετικέ αναλλακτικέ λύσει για τον τρόπο οργάνωση τη λειτουργία και ε, διαφορές. Δεν είναι σαφέ δηλαδή το πώς οργανώνεται και η Eurojust μέσα από τη συνθήκη. Πράγμα το οποίο οδηγεί βέβαια σε συζητήσεις αταρμονούς διαλόγους μεταξύ των διαφορών φορέων, πράγμα το οποίο, όπως είπα, ε, μας επαναφέρει στην ανάγκη να συζητήσουν μεταξύ τους και να λύσουν τα προβλήματα αυτές οι αρχές. Ο κύριος Ντάιρτσι, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Μία παρατήρηση μόνος προς το περιεχόμενος προς την ουσία. Για να εξηγήσω την ασάφεια και απουσία συνενέσεως για την οποία ε, εκφράσατε η μαρτυρία σας και είναι κατανοητή βεβαίως. Απλώς πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι καινούριο πεδίο αρμοδιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Τα τελευταία μόλις χρόνια εμφανίστηκε αυτός ο χώρος και μετακύλησε από τον τρίτο πυλώνα στην ε, νομοθεσία την εσωτερική των κρατών μελών πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Και άρα είναι ασαφές για τα κράτη-μέλη και το πώς θα πρέπει να κινηθούν στον τομέα αυτό, πράγμα που εξηγεί και την ασάφεια και τις διαφωνίες, αν και... Είναι ασαφές το άρθρο της συνθήκης. Πιστεύω ότι εσκεμένα δείχνει μια τάση από τη Eurojust σε, μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή. Και είναι εσκεμένα ασαφές το άρθρο έτσι ώστε να μπορέσει ο κάθε ένας χρόνο να βρει τις λύσεις που του αρμόζουν καλύτερα. Και συμφωνώ σε αυτό που είπατε ότι οι εθνικοί εισαγγελείς θα πούν ότι ναι μπορεί να υπάρχει Eurojust ήδη αλλά εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την ενισχυμένη, την ε, ενισχυμένη εντατική ε, διεθνική συνεργασία δηλαδή μεταξύ των εθνικών αρχών. Ε, παρότι όπως είπαμε υπάρχει ήδη Eurojust αλλά αυτό οφείλεται στο ότι είναι ασαφής η σχετική διάταξη, οι σχετικές διατάξει και είμαστε σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτό που θα βλέπαμε σε ένα σούπερ μάρκετ, ότι μπορεί κανείς να διαλέξει δηλαδή τη λύση που τον βολεύει καλύτερα. Δεν ε, είναι ζηλευτή η θέση της Επιτροπής, δεν θα είναι εύκολο δηλαδή να εξασφαλίσει η πλειοψηφία στο Συμβούλιο προς τη μία ή την άλλη λύση και υπάρχουν κάποιοι που δεν θα υποστηρίξουν καθόλου τη λύση ενός, μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής πέραν των ε, διατυπώσεων τη ίδρυσης της όταν έρθει η στιγμή να Υπάρχουν κάποιοι που είναι την ιδέα την ίδια πάση περιπτώσει πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις και εσείς βέβαια να διαμορφώσετε μια σαφή εικόνα σε σχέση με αυτές τις εναλλακτικέ. Και πιστεύω ότι η έκθεσή μας αυτή τη δουλειά κάνει. Η μελέτη μας σαν στόχο έχει να σας δώσει τις εναλλακτικέ και να σας αφήσει το περιθώριο της επιλογής. Εντάξει κυρία Γιάλα Σέντερ, ικανοποιημένη. Πήρατε τις πληροφορίες που θέλατε. Ναι. Ωραία. Τώρα για σας ο πρόεδρος Νταματζίστρης έχει αναμειχθεί πολύ στη μελέτη αυτή και είχε ενδιαφερθεί μια που ήταν και αυτός δικαστής. Ε, φαντάζομαι έχει μεταφραστεί και στα Ιταλικά για να ενημερωθεί και εκείνο. Είναι άρρωστος δυστυχώς τώρα, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Πάντως το γραφείο του είναι πολύ κοντά εδώ. Οπότε σέρθετε σε επαφή μαζί του και ενημερώστε τον ε, παρακαλώ να δείτε πώς μπορείτε να συναντηθείτε ώστε και εκείνο να βοηθήσει το δικό σας έργο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε κλείνει αυτό το σημείο που ήταν το σημείο 4 και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 5 και που είναι η έκθεση της συναδέλφου Μαρινέσκου. Κοιτάξτε κυρία Μαρινέσκου. Α, μας έχουν έρθει εδώ οι Ρουμάνοι διερμηνείς λέει ο πρόεδρος. Οπότε, ωραία. Γιατί υπήρχε πριν ένα πρόβλημα με τα ρουμανικά στην αρχή. Δεν είχαμε ρουμανικά, βλέπετε, στη συνεδρίασή μας. Τώρα όμως έχουμε. Είχε γίνει κάποια παρεξήγηση ανάμεσα στη γραμματεία μας και τους διερμηνείς, αλλά οι διερμηνείς φρόντισαν πάρα πολύ γρήγορα και έτσι έχουμε τώρα την ε, ρουμανική διερμηνία, οπότε μπορείτε να μιλήσετε ρουμανικά αν θέλετε. Είσαστε εισηγητής κύριε Μαρινέσκου, οπότε σας ακούμε. Παρακαλώ. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πέντε χρόνια υπάρχουν τα ρουμανικά εδώ, οπότε βρίσκω φυσιολογικό να είναι εδώ και η γλώσσα μου, παρόλο που καταλαβαίνω. Λοιπόν, Συνεχίζει στα ρουμανικά ο κ. Μαρινέσκου. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών στο διάφορα κράτη-μέλη. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι φυσιολογικό αυτό, διότι πρόκειται για ένα ποσό που είναι περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Ένα ποσό που έχει δοθεί για τη δραστηριότητα αυτή του παροπλισμού. Η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ορθή τα κράτη-μέλη πρέπει όντως να στηρίζονται στη δράση τους αυτή. Δυστυχώς όμως, από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση και ακόμα και μετά τα πρώτα σχέδια κλεισίματος πυρηνικών αντιδραστήρων δεν ετέθη προθεσμία ούτε για το κλείσιμο ούτε για τα κονδύλια. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο σχέδιο για τον παροπλισμό των πυρηνικών αυτών αντιδραστήρων. Το 2011 και το 2012 θα συζητήσουμε για τον προπολογισμό του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έπειτα έχουμε εξοδέψει πολλά χρήματα για την ενέργεια. Συνεπώς θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε δώσει και για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά πολλές χώρες ξόδεψαν πάρα πολλά για την ενέργεια και πάρα πολύ λίγα για τις δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο και στον παροπλισμό των πυρηνικών αντιδραστήρων. Η συζήτηση αυτή γίνεται σε μια καλή στιγμή πιστεύω. Ε, σύντομα θα δημοσιευθεί έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα τρία σχέδια και το Μάιο ή τον Ιούνιο θα έχουμε την ε, ελεκτική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου δηλαδή. Πρόκειται για έναν έλεγχο επιδόσεων για τις τρεις χώρες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ζητήσουμε από την Επιτροπή και από το ελεγκτικό συνέδριο να μας πούνε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Οι κύριες πτυχές τι δηλαδή πρέπει να πετήσουμε. Ένα, καθορισμό προθεσμίας προκειμένου να δοθούν κονδύλια για τα τρία αυτά σχέδια. Δεύτερον, τη δημιουργία συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα συντονισμού. Η εμπειρία μας λοιπόν είναι ότι τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τα σχέδια για ένα πυρηνικό αντιδραστήρα δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των ε, δύο άλλων περιπτώσεων. Άρα δεν μειώνονται τα ποσά. Θέλουμε λεπτομέρειες για τα σχέδια κλεισίματος επίσης των πυρηνικών αντιδραστήρων. Και αυτό λείπει. Ευχαριστώ πολύ. Eh, eh, Ευχαριστούμε. Πάλι στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κίρχνερ είναι εδώ, έτσι, από τη Γενική Διευθυνσία Ενέργειας. Είναι σημαντικός μάλιστα, πολύ σημαντικός για αυτό το θέμα, γιατί είναι επικεφαλής του, της μονάδας που ασχολείται με τον παροπλισμό πυρηνικών αντιδραστήρων. Οπότε σας δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Μαρινέσκου για την πολύτιμη αυτή έκθεση και ιδιαίτερος για την αξιολόγηση την οποία προέβη τη αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Τις δύο έννοιες τις έχει εντάξει στο πλαίσιο ε, της έκθεσης του με πολύ σαφή τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το στοιχείο. Εν γέννη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τα πορίσματα της έκθεσης. Η Επιτροπή τελεί εν πλήρη γνώση των ζητημάτων που χρήζουν βελτιώσεως και Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία και διαβουλεύση με τα τρία εμπλεκόμενα κράτη-μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουμε βελτίωση και προόδο στα ζητήματα αυτά. Η έκθεση, όπως σωστά αναφέρει ο κ. Μαρινέσκου, έρχεται σε μια πολύ έφετη στιγμή και θα συμβάλλει τα μάλα στην ε, δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το ε, τη συζήτηση του μέλλοντος για την περίοδο μετά το 2013. Και, στην, ε, και συγκεκριμένα για να σας δώσω κάποια παραδείγματα που επισημαίνει και η έκθεσή σας, η υπαγωγή σε όρους ενός ε, λεπτομερούς σχεδίου παροπλισμού και πλήρους αξιολόγησης κόστους και αποτελέσματος καθώς και χρηματο... οικονομικού σχεδίου τι δηλαδή χρειάζεται για να προχωρήσουμε στον παρεπλισμό και από πού θα βρούμε τα κονδύλια που απαιτούνται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται από την έκθεση πολλέ φορέ, σε διάφορα σημεία τη έκθεση, να ενημερώνει, να διευκρινίζει. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη σα για να προσφέρει τι υπηρεσίε αυτέ, τι ε, πληροφορίε αυτέ. Απλώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω, γιατί το θέμα ετέθηκε εχθέ κατά τη συζήτηση γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ήτρε, πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως κύρια προτεραιότητα την τον ασφαλή παροπλισμό. Ευχαριστώ και πάλι για τη σημαντική αυτή έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιβάνοβα. Έχεις δει στο λόγο κανένας άλλος. Και μετά ο κύριος Μαρινέσκου βέβαια μπορεί να πάρει και πάλι το λόγο για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ κύριε Ιβανόβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική του δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης για την οικονομική ενίσχυση και για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς ο παροπλισμός στο Κοσλοντούι στην Βουλγαρία δεν θα ήταν κάτι εφικτό. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα και μετά θέλω να ρωτήσω και κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην παράγραφο 28 που ανέφερε και η Επιτροπή γίνεται κάποια υπόνοια όσον αφορά την ασφάλεια. Η παράγραφος 28 υπογραμμίζει ότι ο κύριος στόχος του παροπλισμού μακροπρόθεσμα των αντιδραστήρων ήταν η ασφάλεια. Εδώ όμως θέλω να ζητήσω να πείτε πιο συγκεκριμένα σε ποια χώρα αναφέρεστε εδώ και σε ποιον αντιδραστήρα. Γιατί τουλάχιστον για την Βουλγαρία οι διάφορες πραγματογνωμοσύνες που έγιναν ε, κατέληξαν στο ότι οι προδιαγραφές ασφάλειας καλύπτονταν. Έπειτα, δεύτερο θέμα. Ε, για τα ποσά που πάνε στον παροπλισμό. Βάσει του κανονισμού τον Ιούλιο του 2010 ήταν ένας κανονισμός που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση στο βουλγαρικό πυρηνικό αντιδραστήρα. Από ό,τι βλέπω εδώ, τα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν βάσει του άρθρου 2 και για άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με το κλείσιμο και τον παροπλισμό των ε, πυρηνικών αντιδραστήρων. Οπότε τα μέσα που διατέθηκαν δεν ήταν αρνητικά όσον αφορά τον ενεργειακό απολογισμό στη Βουλγαρία, διότι πολλά από τα ποσά αυτά χρησιμοποιήθηκαν γενικά για την ενέργεια προκειμένου να αντισταθμίσουμε την απώλεια ενεργειακής ισχύως που είχαμε στη Βουλγαρία. Τέλος, θέλω να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην παράγραφο 25 λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσκολεύεται να πάρει πληροφορίες κατά τη διάρκεια του έργου της. Μπορείτε παρακαλώ να διευκρινίσετε ε, σε ποια χώρα αναφέρεστε, με ποια χώρα έχετε δυσκολίες για να σας βοηθήσουμε δηλαδή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Βάνοβα. Πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις της. Παρακαλώ κύριε Κίχνερ, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Okay, uh, Ναι, βεβαίως. Όταν μιλώ για ασφαλή παροπλισμό, παραπέμπω στο ρόλο μας ε, για την εξασφάλιση υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον, παρα... στον παραπλισμό των τριών αντιδραστήρων, Κοσλοντούι, Ιγναλίνα και Μπουγούνιτσα και τα ζητήματα που προκύπτουν εν ώψη του παραπλισμού αυτού. Είναι το ζήτημα της ασφάλειας πολύ σημαντικό. Κίνδυνος υπάρχει πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με αδιάθετο πυρηνικό ε, υλικό, πυρηνικό καύσιμο δηλαδή, ή με τα απόβλητα τα πυρηνικά και βέβαια υπάρχουν στήματα και προστασία στι δημοσιονομικέ και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ο παροπλισμός πρέπει οπωσδήποτε να είναι ασφαλής και αυτό είναι ο γνώμονος με βάση τον οποίο οργανώνουμε τη δουλειά μας. Για τον κανονισμό στον οποίο αναφερθήκατε, είπατε ότι τα κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί για, την, για τον παροπλισμό και άλλα σχέδια. Ε, ναι, βεβαίως έχουν χρησιμοποιήσει τον παροπλισμό, αλλά και για την ε, ε, λήψη μέτρων περιορισμού των συνεπειών του πρόωρου παροπλισμού. Συμφωνούμε δηλαδή στο να διατεθούν τα κονδύλια στο στόχο αυτών και, τον, και το υποστηρίζουμε. Αυτό άλλωστε έχει ενταχθεί και στις δημοσιονομικές προοπτικές για τη Βουλγαρία για το 2013. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που εντοπίζονται στην έκθεση, που όμως δεν έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα στήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά με κάποιες ανταλλαγές που είχαμε με τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, δηλαδή με τη δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, για τη διαχείριση των σχετικών δημοσιονομικών πόρων. Είχαμε θέσει κάποια ζητήματα με ερωτηματολόγιο, δεν λάβαμε εγκαίρω απαντήσει. Το πρόβλημα όμω επελήθη σύντομα και διμερός με τη βουλγαρική κυβέρνηση τη εποχή και ω εκ τούτου από πλευρά μα δεν μένει κανένα εκρεμέ ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα πλέον δηλαδή ε, ενημέρωσης στοιχείων που είχαμε στήσει. Δεν νομίζω ότι η κυρία Ιβανόβα ικανοποιήθηκε πλήρω, οπότε θα παρέμβει και πάλι. Παρακαλώ κυρία Ιβανόβα. Όχι, ικανοποιήθηκα πρόεδρε από την απάντηση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ τον εκπρόσωπό της. Μία διευκρίνηση έχω να κάνω όσον αφορά το πρώτο θέμα. Δεν πρόκειται για την ασφάλεια του παροπλισμού. Εγώ μιλούσα για το ότι το κλείσιμο φαινόταν ε, εδώ ότι έλεγε ότι έγινε επειδή δεν ήταν ασφαλής ο παιδικός αντιδραστήρας και όχι ότι πρόκειτο για την ασφάλεια παροπλισμού. Και οι πραγματογνωμοσύνες που είχαν γίνει έδειχναν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας με τον ε, πυρηνικό αντιδραστήρα. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση αυτή. Ο πρόσωπος της Επιτροπής, όχι. Ο εισηγητής μήπως για να κλείσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την παράγραφο 28 λέει ότι στόχος της οικονομικής στήριξης ήταν η διασφάλιση ε, των ε, προδιαγραφών ασφάλειας. Πάνω σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε, αυτό πρέπει να τονίσουμε. Με την ένταξη οι τρεις χώρες αναγκάστηκαν να κλείσουν τους πυρηνικούς τους αντιδραστήρες προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της και θα ήταν καλό εφόσον η Επιτροπή ολοκλήρωνε την αξιολόγηση που αναφέρεται εδώ, γιατί έτσι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ενημερωθεί για την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια αξιολόγηση, μια μελέτη που μας ενδιαφέρει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας κύριε Σιγητά. Οι συνάδελφοι έχουν χρόνο να τροποποιήσουν αν θέλουν την έκθεσή σας μέχρι την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Και μετά θα ψηφίσουμε την έκθεσή σας στις 3 Μαρτίου. Έτσι. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Οπότε τελειώσαμε και με το σημείο 5 και ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Σημείο 6. Διάφορα. Υπάρχουν διάφορα. Παρακαλώ. Όχι. Καλώς. Τότε κλείνει η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 10 Φεβρουαρίου. Πέμπτη πριν από το Στρασβούργο δηλαδή. Και έχουμε μπόλικα πράγματα στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συνεργασία. Και καλή επιστροφή για αυτούς που θα επιστρέψουν ε, στις χώρες τους. Ευχαριστώ.